Επίτροπο απαντησει απαντήσει αρχής πινκ-πονγκ, δηλαδή ε, ερώτηση-απάντηση και ούτω καθεξή. Θα ξεκινήσουμε με ένα γύρο ερωτήσεων από του επικεφαλεί των 7 πολιτικών ομάδων προ την Επίτροπο. Και ο καθένα θα έχει 7 λεπτά, 1 λεπτό για ερώτηση, 2 λεπτά απάντηση, δύο λεπτά συμπληρωματική ερώτηση, ένα λεπτό απάντηση. Στο δεύτερο γύρο θα υπάρξουν 38 ερωτήσεις με ναι, τρία λεπτά ε, κάθε μία, δύο λεπτά για την ερώτηση και ένα λεπτό για την απάντηση. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον κύριο Λεμπρούν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Περιφερειών, για μια σύντομη δήλωση. Στο τέλος, η κυρία Κορίνα Κρέτσου, υποψηφία επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, θα έχει πέντε λεπτά, χρονοφυρίδα πέντε λεπτών για τις ε, καταληκτικές της παρατηρήσεις. Ο καταμερισμός του χρόνου αγόρευσης ακολουθεί τη μέθοδο DONT, βάσει του οποίου η, τάξη, η σειρά των παρεμβάσεων έχει αποφασιστεί από τις πολιτικές ομάδες. Οι ερωτήσεις δεν, είναι, ε, δεν κατηγοριοποιούνται αναθέματα. Ε, θα πρέπει να τονίσω ότι είναι ουσιαστικό όλοι οι ομιλητές να τηρήσουν τα χρονικά όρια για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, γιατί αν όχι δεν θα έχουμε, θα ξεπεράσουμε το χρόνο μας και ορισμένα μέλη δεν θα έχουν δυνατότητα να πάρουν το λόγο. Ακριβώς όπως στην Ολομέλεια, ένα ρολόι θα, θα δείχνει πόση ώρα έχετε μιλήσει. Έχουμε διερμηνία στις 23 γλώσσες. Όλοι οι μιλητές μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα τους, αλλά παρακαλώ να μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Και τώρα μετά από αυτές τις παρατηρήσεις Ελπίζω ότι η διαδικασία είναι ξεκάθαρη για όλους και ε, θα κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασης και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην υποψηφία επίτροπο για μια παρουσίαση η οποία δεν θα ξεπεράσει τα 15 λεπτά. Αυτή η παρουσίαση θα ακολουθεί από χρόνο υποβολής ερωτήσεων και απαντήσεων